πολίτε μα μα ζητούν να αναλάβουμε δράση για να σταματήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη, να σταματήσουμε την αποψήλωση των δασών, να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν πρόκειται να επιβραδυνθεί λόγω μεμονωμένων δράσεων, γιατί δεν γνωρίζει σύνορα από την Κίνα στι Ηνωμένε Πολιτείε, από την Αυστραλία, από πάρα πολλέ ε, περιοχέ του κόσμου μα επηρεάζει αυτή τη στιγμή η κλιματική αλλαγή και μπορούμε να νικήσουμε μόνο αν συνεργαστούμε από κοινού, δεν αφήσουμε κανέναν εκτό. Θα πρέπει να λάβουμε δράση για τον άνθρακα, για τι φροντικέ απαλλαγέ ε, στον τομέα τη αεροναυτιλία. Τα ροκτικά καύσιμα ανήκουν στο παρελθόν. Θα πρέπει να τανίσουμε το μέλλον τη ενέργεια. Α εγκαταλείψουμε τι παλιέ τεχνολογίε, α δημιουργήσουμε και σχηματοδοτήσουμε νέε. Α δώσουμε νέα όθηση στην Ευρώπη, α επενδύσουμε περισσότερο στην επιστήμη και την καινοτομία. Α συνάψουμε εμπορικέ συμφωνίε οι οποίε συμμορφώνουν συμμορφώνονται με τη Συμφωνία των Παρισίων. Έχουμε λοιπόν την ακόλουθη επιλογή ή από κοινού θα συνεργαστούμε και θα μας αλλάξει το ίδιο το κλίμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενος ο συνάδελφος Πέρνσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε έχουμε εξαιρετική ευθύνη έναντι των επόμενων γενναιών, έναντι των παιδιών μας. Πρέπει να τους δώσουμε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι βιώσιμος, πιο καθαρός, πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε αυτό το επίπεδο, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια στρατηγική, να είμαστε ανεξάρτητοι από την Ρωσία και τη Μέση Ανατολή ως προς τον εφοδιασμό ενέργειας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε στην Ευρώπη, τι είδους αηφόρο ενέργεια μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και τρίτον, χρειαζόμαστε πιο ισχυρές οικονομίες ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να δώσουν ένα καλό μέλλον στα δικά τους παιδιά. Χρειαζόμαστε μια ειλικρινή μετάβαση για τους πολίτες, για τη βιομηχανία μας. Ε, έχουμε για παράδειγμα την υποδομή του αερίου η οποία μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για πιο βιώσιμους ε, στόχους. Και πρέπει ταυτόχρονα να ε, μεριμνήσουμε ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος ε, στην οποία θα υπάρχει όφελος και κέρδος. Όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός ε, και οι διαστάσεις είναι τέτοιες που πρέπει να δράσουμε αμέσως. Η γεωργία είναι κυρίως αυτή που πλήττεται από την αλλαγή του κλίματος σε σχέση με άλλους τομείς ταυτόχρονα οι γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι βασικοί θεματοφύλακες ε, του περιβάλλοντος. Η γεωργία, οι αγροτικές περιοχές ε, ε, είναι υπεύθυνοι για την ευημερία των ανθρώπων και για την ποιοτική διατροφή τους. Ε, λένε ότι στα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί κατά 30% ο πληθυσμός. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ε, θα είμαστε αυτοί που θα αναλάβουμε το, το ρόλο του πιο σημαντικού παραγωγού τροφίμων. Ε, ο κίνδυνος λοιπόν της αλλαγής του κλίματος είναι μεγάλος και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για μια οικολογική γεωργία η οποία θα είναι καλή και ε, για το κλίμα και για το περιβάλλον. Ε, συνάδελφο την Μπενχουμέα, Μπενχουμέα. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το περιβάλλον και η βιωσιμότητα είναι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε τις φυσικές καταστροφές, τις θεομηνίες. Για παράδειγμα, οι πλημμύρες που είχαμε στην Ισπανία το Σεπτέμβριο, όπου δυστυχώς είχαμε και θύματα. Αλλά δυστυχώς η αριστερά εδώ και πολλά χρόνια θεωρεί ότι η συζήτηση είναι μόνο δική της. Η αριστερά προσπαθεί να έχει αποκλειστικά κάθε πρόταση και να κάνει τη συζήτηση με τέτοιου όρου που να μην ε, προ, ε, προ, προτείνονται ρεαλιστικέ λύσει. Για παράδειγμα, τα χρησιμοποιεί για να κατηγορήσει ε, τον καπιταλισμό και την παγκοσμιοποίηση. Αυτό τους έχει μείνει από την τρομερή του ήττα το 1989. Η πρόοδος και η ανάπτυξη δεν είναι εχθροί του περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε τον τεράστιο ρόλο που παίζει ιδιωτική πρωτοβουλία για την προστασία των οικοσυστημάτων παντού στην Ευρώπη και περιοχών φυσικού κάλους. Πρέπει να ασχοληθούμε με το άτομο, με το τοπικό περιβάλλον, την ατομική ευθύνη και την τοπική αυτοδιοίκηση. Να σταματήσουμε λοιπόν να αξιοποιούμε το περιβάλλον ως πρόσχημα για να κάνουμε άλλες μάχες. Να ξεφύγουμε τις υπερβολές και τις κατηγορίες για να βοηθήσουμε πραγματικά τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια. Βίρκουνεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, προκειμένου να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε, αλλά μην ξεχνάμε τι έχουμε ήδη επιτύχει. Οι στόχοι για το 2020 θα επιτευχθούν και θα τους ξεπεράσουμε μάλιστα. Και μέχρι το 2030 έχουμε έναν φιλόδοξο στόχο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι και οι στόχοι αυτοί για το 2030 θα επιτευχθούν και μάλιστα θα τους ξεπεράσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις και μην ξεχνάμε ότι έχουμε εγκρίνει και πάρα πολλού κανονισμού. Έχουμε ήδη μία δέσμη καθαρή ενέργεια, μία οδηγία όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, νέου περιορισμού όσον αφορά τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, ιδίω για τα βαρέα οχήματα. Έχουμε μια στρατηγική για τα πλαστικά. Έχουμε απαγορεύσει την χρήση πλαστικών μίας χρήσης. Πολλές θετικές αποφάσεις λοιπόν έχουμε πάρει στο παρελθόν. Τώρα θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη θετική δυναμική και θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο του 55% μέχρι το 2030. Περισσότερες χώρες μπορούν το να το πετύχουν αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ σημαντικούς φιλόδοξους ηγέτες όσον αφορά την περιβαλλοντική αυτή πολιτική. Ο κύριος Καρβάλιο, η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και όλη η συζήτηση δεν είναι συζήτηση πολιτικής φύσης έχουμε συγκεκριμένες αποδείξεις ενώπιόν μας που μας καλούν να αναλάβουμε δράση με ευθύνη και φιλοδοξία χωρίς να δίνουμε φρούδες ελπίδες ε, στους πολίτες, χωρίς να δίνουμε κενές υποσχέσεις τις οποίες δεν πρόκειται να ελοπίσουμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε εφαρμόζοντας τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει και ας χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες. Δυστυχώς πολλές από αυτές δεν υλοποιούνται ακόμα στην πράξη, αλλά πρέπει να πάμε και λίγο πιο μακριά, να αναλάβουμε δηλαδή επιπλέον μέτρα, αλλά πάντα αφού κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση του αντικτύπου τους. Για να προχωρήσουμε όμως περαιτέρω χρειάζεται περαιτέρω επιστημονική έρευνα, καινοτομία, περισσο... μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα τη τεχνολογία. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συμφιλιώσουμε τη φιλοδοξία τη καταπολέμηση κλιματική αλλαγή με μια σημαντική ηγεσία στον τομέα της βιομηχανίας που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τον τρόπο ζωής μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα, κάρτα όμως δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Ο επόμενος είναι Άλφος Κέλλη. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο στην Συμφωνία του Παρισιού στο Μαρακές και πέρυσι στην Πολωνία και ήμουν και εισηγητής ε, ε, σε αυτή τη συζήτηση ε, και τα, βλέπω ότι τα πράγματα τώρα κινούνται. Έχουμε μια οικολογική εκτακτή ανάγκη. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να δρουν. Ε, έτσι λοιπόν χαιρετίζω τη δέσμευση της ε, κληγμένης πρόεδρου Φοντερ Λάιεν για την ε, Πράσινη Συμφωνία, μια πρόταση που θα μπει τις πρώτες 100 μέρες. Είναι ζωτική σημασία σε όλα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε ως εκτακτή ανάγκη. Το είπαμε αυτό όταν είπαμε ότι οι στόχοι πρέπει να ανέβουν προς τα πάνω. Είναι καλό αυτό, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να ξεχνάμε αυτούς ε, που θα επηρεαστούν. Πρέπει να είναι δίκαιη η μετάβαση. Είναι ζωτική σημασία και πρέπει να λογοδοτούν τα κράτη κάθε χρόνο για να βλέπουμε πώς θα προοδεύουν. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την εκτακτή ανάγκη και θα έχουμε διασφαλίσει το μέλλον των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ε, τελευταία συνάδελφος, ο συνάδελφος Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό εδώ το σώμα πάντα όταν μιλάμε για ψηφίσματα και για το κλίμα είναι πάντοτε έτσι ιδιαίτερα εκφραστικό. Όμως ε, το πρόγραμμα ε, είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν άδειες ε, για ρήπανση, ενθαρρύνονται οι μία ή φόρες μορφές κατανάλωσης, ε, ευνοούνται η φορες μορφες καταναλωσης βνοουνται παραγωγή και μια γεωργία που είναι υπέρ της agribusiness και κατακαιρματίζει την μικρή γεωργία τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε τεράστιες ε, πόλεις. Ε, το πρόβλημα είναι ο προϋπολογισμός, οι πόροι που δίνονται ε, τελικά για τα όπλα και όχι για την περιφερειακή συνοχή. Θα πρέπει λοιπόν εδώ όχι απλώς να επαναλαμβάνουμε δηλώσεις, πρέπει τελικά πολύ σοβαρά να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντιφάσεις. Και τώρα έχει το λόγο ο Επίτροπος Έτιγκερ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, μαζί με τον συνάδελφό μου εδώ έχω συζητήσει και έχω σημειώσει τα ε, πολυάριθμα σχόλια που κάνατε για την γεωργία, την βιομηχανία, για τους πολίτες, για τα κτίρια για την οικονομία μας. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα που διαφαίνεται και να πω ότι θέλετε να σκίσετε πίεση ώστε να ε, ορίσουμε συγκεκριμένα αυτά που προσδοκάτε μέσα στα πλαίσια της νέας ε, Κομισιόν και μέσα από τις πρώτες 100 ε, μέρες όπου θα κατατεθούν νομοθετήματα μέσα στα πλαίσια του πράσινου πακέτου και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με εταίρους εκτός της Ευρώπης. Όλα αυτά θα πρέπει να επιταχυνθούν και έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών και να δείξουμε πόσο έκτακτη είναι αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι η συζήτηση ήρθε σε ένα σωστό σημείο. Είμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή στα μέσα μιας διαβούλευσης για τον ε, προϋπολογισμό, άρα ε, μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις. Υπάρχει το Transition Fund, ε, ε, υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι μηχανισμοί που αυτή τη στιγμή συζητούνται από τους εισηγητές της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ο συνάδελφος Τίμερμαν, θα μάθει για όλα αυτά που μου είπατε από μένα και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ εκ μέρους ε, του ε, Συμβουλίου η Υπουργό κυρία Ράιναν, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Άκουσα προσεκτικά τις παρεμβάσεις, τις προτάσεις σας και σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα στην αρχή της συζήτησης, ε, το να κλιμακώσουμε τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής είναι τώρα μια έκτακτη ανάγκη. Πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα, να δείξουμε ηγεσία, ηγετική διάθεση, να δράσουμε ως ηγέτες ε, και η Προεδρία μας εργάζεται σκληρά ώστε να πετύχουμε αυτή τη θέση. Επίσης, στοχεύουμε σε μία συμφωνία ε, για την στρατηγική τη ουδετερότητα σε επίπεδο εκπομπών του του άνθρακα. Ελπίζουμε ότι τον Δεκέμβρη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε θετικά βήματα. Θα είναι τεράστιο επίτευγμα αν όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050 καταφέρουμε να είμαστε ουδέτεροι κλιματικά. Τώρα, όσο πιο γρήγορα ε, αναλάβει καθήκοντα η νέα Επιτροπή και όσο πιο γρήγορα κατατεθεί η πρόταση για το, δίκαιο, ταμείο, ε, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ε, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να βάλουμε αυτά τα σημεία στον μελλοντικό προϋπολογισμό, στο ΠΔΠ γιατί πραγματικά η δίκαιη μετάβαση είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε το θέμα του κλίματος. Είναι αλήθεια ότι αυτό το θέμα ε, επιζητά μια ευρεία και προσεκτική συζήτηση. Όσο πιο πολύ συζητάμε, τόσο πιο καλά μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον. Η Προεδρία μας έχει το σύνθημα «Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για μια βιώσιμη Ευρώπη και ένα βιώσιμο μέλλον». Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ε, με αυτό τελειώνει η συζήτηση για το ε, θέμα αυτό και πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η συζήτηση για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, καλουσιάζω εδώ τον Κλάους Χάινερ Λένε, τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου ε, σύμφωνα με το νέο σύστημα, ε, οι μπλε κάρτες ε, και η αυθόρμητη ζήτηση του λόγου γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Αν θέλετε λοιπόν να μιλήσετε, θα πρέπει να το κάνετε από τώρα. Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι το τέλος της συζήτησης. αν όλοι έχουν κάτσει στις θέσεις τους. Nehmen sich die Zeit, die Sie Helena. Παρακαλώ πάρτε το χρόνο που χρειάζεται. Θα περιμένουμε να φύγουν οι επισκέπτε μα από το Συμβούλιο και θα πάρει το λόγο ο κύριο Λένε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, κύριε εκπρόσωποι τη Προεδρία, κύριε Επίτροπε κυρίε και κύριοι, χαίρομαι πολύ που σήμερα μαζί με τον ε, κύριο Λάζαρο Λαζάρου, τον ε, διακεκριμένο συναδελφό μου, συναδελφό μου μπορώ να σα παρουσιάσω την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Για τη διαδικασία απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου με την ε, έκθεση για τον προπολογισμό του 18. Γιατί πρόκειται. Θέλω να σε ενημερώσω για την διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης. Πώς έχει τώρα. Στην ετήσια έκθεσή μας ασχολούμαστε με την δήλωση αξιοπιστίας. Εάν δηλαδή οι πόροι που εσείς ε, αποφασίσατε πέρυσι δαπανήθηκαν σωστά. Τυπικά σωστά και αν βοήθησαν την οικονομία μας. Έχουμε τους ονοποιημένους λογαριασμούς για το 2018, τους οποίους ελέγξαμε. Κατά την ε, κρίση μας η κατάσταση των οικονομικών της Ένωσης είναι καλή και δεν υπάρχουν σοβαρά σφάλματα. Δηλαδή, εγκρίναμε χωρίς επιφυλάξεις ε, τον απολογισμό. Και δεν θεωρούμε ότι το ποσοστό σφαλμάτων είναι ουσιώδες για τα έσοδα. Για τις δαπάνες θεωρούμε ότι είναι 2,6%. Αυτό σημαίνει ότι κατά τις εκτιμήσεις μας 2,6% των πληρωμών δεν θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό γιατί δεν ε, συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο για τη δαπάνησή τους. Αλλά υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση. Ο τρόπος πληρωμών των ευρωπαϊκών πόρων έχει μεγάλες επιπτώσεις στο κίνδυνο σφάλματος. Για τις δαπάνες είναι πολύ περίπλοκες οι διατάξεις. Για τον μισό περίπου προπολογισμό που είναι αποζημιώσεις όπως λέγονται. Δηλαδή, επιστρέφονται αποζημιώσεις για το κόστος που έχει ε, προκύψει στην έρευνα, για την απασχόληση, για την ανάπτυξη της υπαίθρου, την ανάπτυξη των φτωχότερων κρατών. Ενώ για τις λεγόμενες πληρωμές ε, μέσω απαιτήσεων έχουμε πολύ χαμηλότερο ποσοστό σφαλμάτων. Εδώ οι δικαιούχοι πληρώνονται εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, άμεσε επιδοτήσεις στη γεωργία, διοικητικέ δαπάνες, υποτροφίες για σπουδαστέ ή η βοήθεια που δίνουμε από τον προπολογισμό σε τρίτες χώρες. Δηλαδή, γύρω στο 50% των ελέγχων που κάναμε δεν ε, ανέδειξαν ουσιώδες ποσοστό σφαλμάτων. Οπότε για τρίτη συνεχή χρονιά δώσαμε ανεπιφύλακτη έγκριση, απαλλαγή. Δηλαδή λέμε ναι μεν αλλά. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη διατήρησαν τις προόδους που είχαν σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Οπότε είχαμε και θετικά στοιχεία. Ωστόσο, Υπάρχουν κάποιοι τομείς που μας ανησυχούν γιατί έχουν υψηλό ποσοστό σφαλμάτων. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν περαιτέρω. Στα πλαίσια της πολιτού στρατηγικής, της, στρατηγικής του, το ελεκτικό συνέδριο εξετάζει κατά πόσον η πιστοποίησή του γίνεται με το σωστό τρόπο, με τεστ. Δηλαδή, θέλουμε στο μέλλον να βασίζουμε τις εκτιμήσεις μας σε ε, αξιολογήσει που θα κάνουμε και σε επίπεδο Κομισιών και σε επίπεδο κρατών μελών, αν πρόκειται για μεικτή διαχείριση. Θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε τι αναγκαίε προποθέσει για να σημειωθούν πρόοδοι σε αυτή τη νέα μέθοδο αξιολόγηση. Και θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία, κύριε Επίτροπε Έτιγα, για να σα ευχαριστήσω και εσά και του συνεργάτε σα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία που θα έχουμε με τον διάδοχό σα. Είμαι πεπισμένος ότι θα υπάρξουν ε, διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε περιορισμένα θετικά βήματα ούτως ώστε να επιδιώξουμε να αξιοποιούμε όλοι τις εργασίες που κάνουν οι ΜΕΝ και οι ΔΕ και να αποφεύγουμε έτσι τις επικαλύψεις. Δηλαδή Επιτροπή και Ελεκτικό Συνέδριο. Αξιότιμοι βουλευτές. Εάν εξετάσετε τα απορίσματα και της συστάσεις μας θα δείτε πολύ συγκεκριμένα τι προτείνουμε. Η έκθεση αυτή είναι ε, μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού εξέτασε τα επιμέρους κεφάλαια. Επειδή σαν πολλοί από εσά εκεί, δεν πρόκειται τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Κυρίε και κύριοι, κύριοι βουλευτές, κυρίε και κύριοι βουλευτές, κάτι που θέλω να καταστήσω απόλυτα σαφές. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ξεκινάει μια νέα θητεία, ένα κράτος μέλος είναι σε διαδικασία αποχώρησης και τα άλλα 27 κράτη-μέλη στο τελευταίο τμήμα των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 21-27. Η εργασία ελέγχου που σας ε, παρουσίασα σήμερα καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα για τρίτη συναπτή χρονιά πληρεί τα υψηλά κριτήρια ελέγχου για τη χρήση των δημοσίων πόρων. Από την επόμενη Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη αναμένουμε να συνεχίσουν αυτές τις προσπάθειες και να βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση. Και βασιζόμεθα και σε όλους εσάς. Μαζί πρέπει όλοι να φροντίσουμε να συμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Επίτροπος. Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε Λένε, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Λένε και όλη του την υπηρεσία για μια αξιόλογη εργασία και πολύ δίκαιη συνεργασία που τα τελευταία τρία χρόνια βιώσαμε με την ομάδα μου. Και νομίζω ότι από κοινού κάναμε προόδους ότι, και ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα περισσότερες ε, προόδους εμείς ε, στην Κομισιόν, ε, στον Κέλεγχο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου με την Συμβουλή των Εμπειρογνωμόνων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είμαστε σε υψηλά στάνταρτ σε επίπεδο διαφάνειας. Ε, το παλέψαμε και ως προς την λογοδοσία ε, είμαστε συνεπείς γιατί μιλάμε για τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών μας. Η νέα επιτροπή Λοιπόν, ε, στην Νέα Επιτροπή κληροδοτούμε μια καλή κατάσταση. Για δωδέκατη φορά λοιπόν παίρνουμε μία δήλωση αξιοπιστίας χωρίς επιφυλάξεις. Ε, την τελευταία χρονιά καταφέραμε ε, να έχουμε ένα επίπεδο λαθών 2,6%, 4,7% ε, για πέμπτο έτος επίσης και τρίτον για τρίτη φορά σε σειρά το ελεγκτικό συνέδριο ε, φτάνει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να δώσει αρνητική αλλά μια θετική με επιφελάξεις ε, ε, γνωμοδότηση. Τέλος, μαζί ε, γράψαμε την έκθεση για τα προγράμματα και μπορέσαμε να βελτιώσουμε τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός παίζει σημαντικό ρόλο για εκατομμύρια πολίτες, γεωργούς, επιστήμονες, ερευνητές, ε, επιχειρηματίες, startups ε, και φοιτητές. Τα τρία τέταρτα ε, αυτού του, των δαπανών τα διαχειριζόμαστε από κοινού με τα κράτη-μέλη και αυτή η συνεργασία βασίζεται σε μία αξιολόγηση βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου έτσι ώστε ε, όλοι μας ε, να δρούμε σύμφωνα με αυτό και τα κράτη-μέλη. Επίσης, στην πολιτική συνοχής και στην γεωργική πολιτική όπου πηγαίνει περίπου το 70% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και στο οποίο οφείλονται και οι εθνικές και περιφερειακές ενισχύσεις ε, είναι ε, ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Θέλουμε να έχουμε καλή και αποτελεσματική διαχείριση των ε, των πόρων μας. Θέλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη δομή με ξεκάθαρη καθαρή λογοδοσία για όλους ε, όσους συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι επιπτώσεις των λαθών που ε, προκύπτουν, το λεγότερο error rate, ε, είναι μικρότερη η επίπτωση και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και από τα κράτη μέλη και από τους ωφελούμενους να ζητούμε πίσω λεφτά τα οποία δεν έχουν δοθεί σωστά. Υπάρχουν δύο ε, σημεία. Το σημείο της πληρωμής ε, και το σημείο των διορθώσεων. Το σημαντικός αριθμός είναι ο τελευταίος. Και τα τελευταία χρόνια οι εκτιμήσεις λένε ότι είναι μόνο 0,8%. Αυτό που πληρώνεται στους πολίτες τελικά είναι αυτό το οποίο ε, με όλες αυτές τις προσπάθειες δεν υποπίπτει σε λάθη τα τελευταία έτος επίσης ε, καταφέραμε να ε, αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα στη διαχείριση των προγραμμάτων συνοχής σε κάποια κράτη-μέλη. Και εδώ και μόνο εδώ, στο 28 κράτη, είχαμε περισσότερα λάθη από ότι, σφάλματα από ότι στο παρελθόν, το προηγούμενο έτος. Και προσπαθήσαμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τη Συμβουλή μας, ε, με την ε, ε, απλούστευση του επόμενου σχεδίου του προπολογισμού να λάβουμε μέτρα απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Έγιναν και κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και φάνηκε μέσα από αυτούς ότι υπήρχαν ε, κάποια ασφάλματα τα οποία ε, ε, οφείλονταν σε συγκεκριμένες οικονομικές κουλτούρες. Νομίζω ότι οι περίπλοκες διατάξεις οδηγούν σε λάθη. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η απλούστευση αλλά πρέπει να υπάρχει και μια εκπαίδευση, μια επικοινωνία, έτσι ώστε οι λήπτες, των, οι ωφελούμενοι των ευρωπαϊκών πόρων να έχουν ένα πιο εύκολο έργο. Ε, μετά από το 2020 ζητούμε να υπάρχει περισσότερη απλούστευση και θα ζητήσω και από εσά τους νομοθέτες ε, ε, να έχετε πιο συγκεκριμένες διατάξεις για το πλαίσιο του προϋπολογισμού που θα οδηγήσουν σε αυτή την απλούστευση και δεν θα ανανεώσουν αυτή την ε, περιπλοκότητα που οδηγεί στα λάθη. Ε, σε συνεργασία με τους εταίρους μας ε, θα προσπαθήσουμε να πατάξουμε και τις αιτίε των σφαλμάτων. Ας πάμε τώρα στις επιδόσεις, στην απόδοση. Έχουμε επιτύχει κάποια πράγματα τελευταίο έτος ε, όσα πραγματικά κάνει μια επισκόπηση για το πώς ε, ε, τηρούνται οι προπολογισμοί σε όλο τον κόσμο και πραγματικά είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Εμείς στην έκθεσή μας προσπαθήσαμε με απλό και αναλυτικό τρόπο να δώσουμε πληροφορίες για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και κάναμε πολύ σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι ε, δεν θα έχουμε μόνο μέτρα που οδηγούν στην πρόοδο, αλλά θα βασίζονται και σε συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα στοιχεία που θέλουμε εμείς να πετύχουμε για να κινητοποιηθεί η Ευρώπη. Η Κομισιόν λοιπόν είναι αποφασισμένη ε, σε αυτό το ε, θέμα να βελτιστοποιήσει τις προτεραιότητες της. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα φανεί και στο επόμενο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Θα έχει κεντρικό ρόλο. Θέλουμε απλώς ε, πιο ξεκάθαρες διατυπώσεις ε, που θα είναι στο επίκεντρο του θέματος, έτσι ώστε οι πολίτες μας να λαμβάνουν τις βέλτιστες πληροφορίες ε, για τον προπολογισμό της Ευρώπης. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Λένε και να ε, πω ότι είμαστε ησύχοι για όλη την ομάδα στο Ελεκτικό συνόδριο αλλά και για την Επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο. Όπως είπε και ο προηγούμενος πρόεδρος, θεωρώ ότι η δουλειά που κάνετε εδώ είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και στο στόχο. Ε, ε, νομίζω ότι τον Νοέμβριο ε, στις ακροάσεις καλό θα είναι να συζητήσουμε αυτό το θέμα και όταν έρθει η Επίτροπος για την προπολογισμό σε εσά τον Δεκέμβρη να συζητήσετε το θέμα πιο ενδελεχώς. Σας εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστώ. Επειδή έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, σας παρακαλώ οι επόμενοι ομιλητές να τηρούν το χρόνο τους. Δύο λεπτά για το ΕΛΚ. Κύριε Χολμάη. Κύριε Πρόεδρε Λένε, αγαπητέ κύριε Λαζάρου, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά το Ελεκτικό συνέδριο για τη θαυμάσια συνεργασία. Θαυμάσια πραγματικά. Και για την ποιότητα της εργασίας που μας αποστέλλεται. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο κύριο Έτιγκερ που έχει κάνει πολλέ προτάσεις, ή μάλλον που έχει υιοθετήσει πολλές προτάσεις μας και συγκεκριμένα τις έχει υλοποιήσει. Θα διαπιστώσατε ότι γενικά η τάση, όπως λέει και ο πρόεδρος λένε, είναι θετική. Πολλά θέματα βεβαίως ε, μας δημιουργούν ερωτηματικά για το επόμενο ΠΔΠ. Πρώτον, οι αμοιβέ που βασίζονται σε αποζημιώσεις ή επιστροφές μοιάζει να έχουν υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων. Μήπως έχει να κάνει με το λεγόμενο gold plating, δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη κάνουν ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση από ό,τι θα ήταν αναγκαίο, βάζουν και άλλα κριτήρια, περιπλέκουν τις διαδικασίες. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επόμενο πιδελταπή να ασχοληθεί πολύ με το θέμα απλούστευση και να το συζητήσει σε βάθος με τα κράτη-μέλη. Διότι εάν ε, πληρώνουμε εκεί που δεν θα πρέπει να πληρώνουμε, αυτό έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα. Και τα κράτη-μέλη πολλές φορές βέβαια μεταθέτουν την ευθύνη στην ε, Κομισιόν. Παρά το ότι δεν είναι η Κομισιόν αυτή που εφήβρε αυτές τις διαδικασίες. Δεύτερον, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν δυσχέρειες ε, με την δημόσια διοίκησή τους. Δεν θέλουμε τώρα να δακτυλοδεικτούμε κανένα, αλλά Πρέπει να φροντίσουμε να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να συμπεριλαμβάνονται στη συζήτηση και κατόπιν να συμπεριλαμβάνονται και στον, ε, στη συζήτηση για το καθορισμό των μέτρων και μετά και στον έλεγχο. Να τους δώσουμε τεχνική βοήθεια και στήριξη. Ούτως ώστε να μπορούν να δουν αυτόνομα, να μπορούν να κάνουν καλούς εσωτερικούς ελέγχους και υποβολή ε, ετοιμάτων χρηματοδότησης να περνάει από τις δημόσιες αρχές με το σωστό και διαφανή τρόπο. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Η Πέγκοβα. Πένκοβα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, κύριε Λένε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δήλωση που κάνατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά που περιγράψατε με τόση λεπτομέρεια τα περιεχόμενα της αιτήσει αυτής έκθεσης. Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την τελική αυτή γνωμοδότηση της αιτήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου του 2018. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε κάποιους τομείς βλέπουμε μείωση του ποσοστού σφάλματος. Ωστόσο, βλέπω ότι υπάρχει ένα υψηλότερο ποσοστό σφάλματος, με συγχωρείτε, στον τομέα της συνοχής. Ορισμένα δεδομένα που μας έχουν δώσει οι διευθύνσεις περιφερειακής πολιτικής προκαλούν ανησυχίες και θα πρέπει επ' αυτό να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το βλέπουμε αυτό και στο όλο ψήφισμα το οποίο έχουμε για την απαλλαγή. Θα ήθελα να χαιρετήσω επίσης την πιλωτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πιο στενή του συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Σαστέλη, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για την παρουσίαση τη ετήσια έκθεση, αλλά και για το όλο έργο το οποίο έχει επιτελέσει και αυτό και οι ελεγκτέ του. Και όπω είχα και τη δυνατότητα να πω στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή, πραγματικά με την παρουσίαση αυτή ξεκινάει η διαδικασία απαλλαγή. Βρισκόμαστε λοιπόν στι απαρχέ τη εργασία μα και Σίγουρα το έργο μα δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε ένα προπολογισμό ο οποίο θα είναι φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση θα πρέπει να δώσει υποσχέσει τι οποίε δεν μπορεί επίτα να τηρήσει. Αν τώρα η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι εν γέννη θετική, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια επιμέρου σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε όλο ιδιαιτέρω. Αναφέρομαι αυτή τη στιγμή σε προβλήματα τα οποία δεν είναι νέα. Για παράδειγμα, η εξέταση των κανόνων αποζημίωσης, όπου έχουμε πολύ σημαντικά σφάλματα, το ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις δαπάνες υψηλού κινδύνου, το χαμηλό επίπεδο απορρόφησης σε κάποιες χώρες, το gold plating, αναφέρθηκε από την κυρία Χολμάιρα αυτό, το αίτημα για περαιτέρω διοικητική απλούστευση, το ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να συλλέγουμε περισσότερο του ιδίου πόρου, ιδίω αυτού που προκύπτουν από του δασμού, καθώ επίση και τα σφάλματα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Το λεκτικό συνέδριο μα είπε ότι όλα τα θεσμικά όργανα και όλε οι αρχέ θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να καταφέρουμε να παρακολουθούμε σωστά την εφαρμογή των κανόνων. Ελπίζω λοιπόν ότι και το Ελεκτικό Συνέδριο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πλουστεύσουν του κανόνε του ελεγκτικούς προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία των δεδομένων αλλά και η επίπτωση των πολιτικών μας επιτόπου. Θα πρέπει να έχουμε δημοσιονομικού ελέγχου οι οποίοι να είναι πιο αποτελεσματικοί. Και όπω ξέρετε ο υπολογισμό των επιδόσεων και των επιπτώσεων των επιδόσεων των δημοσιονομικών πραγματικά περνά και από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Θεωρώ λοιπόν ότι το Ελεκτικό Συνέδριο θα πρέπει να μπορεί να αποτιμά, να αξιολογεί και τις επιδόσεις, την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών πολιτικών. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Η κυρία Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας όσον αφορά την τελευταία αυτή έκθεση. Βλέπουμε εδώ πέρα τα οικονομικά δεδομένα όσον αφορά το έτος 2018. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο προπολογισμό μας πρέπει να είναι πάντα βιώσιμος. Οι καθυστερούμενες πληρωμές, οι συσσωρευμένες πληρωμές που δεν έχουν καταβληθεί δεν αναφέρονται μόνο στο 2018, αλλά επηρεάζουν πάρα πολύ και τα πράγματα για το μέλλον. Οι εκρεμείς αυτές δεσμεύσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια χρόνια και το 2018 φτάσαμε σε έναν ιστορικό αριθμό με 281 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία κρεμούν και δεν έχουν καταβληθεί ακόμα ως πληρωμές. Και οι προπτικές δείχνουν ότι αυτό θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και ξέρετε ότι αυτό δεν είναι μόνο μια ανησυχία λογιστικής φύσης αλλά και πολιτικής φύσης. Θα πρέπει οι απαραίτητες πιστώσεις πληρωμών να καλύπτουν όλες τις δαπάνες και κατά τα πρώτα έτη του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου διαφορετικά θα τεθεί εν κινδύνο το ίδιο το πολιτες δημοσιονομικό ε, πλαίσιο και τα επιμέρους προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που ενδεχομένω να αντιμετωπίσουμε λόγω των καθυστερούμενων αυτών πληρωμών ακόμα και διαρθρωτικά προβλήματα. Θα πρέπει να μειωθούν οι μη καταβληθήσει ορευμένε πληρωμέ και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τι χώρε εκείνε που έχουν καθυστερήσει και υπολείπονται και να καταφέρουμε να έχουμε ένα προπολογισμό βιώσιμο όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει επίση επίση να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφηση των κονδυλίων και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω τη απλούστευση. Το αναφέρατε αυτό. Θα πρέπει να αποφύγουμε να ασκήσουμε έντονη πίεση από την αρχή του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Κύριο Κούζ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν δεν υπήρχε το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο, θα έπρεπε να το επινοήσουμε. Η εργασία του κύριε Πρόεδρε, λένε είναι ιδιαίτερο σημαντική για όλους μας. Και το εκτιμούμε. Αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Η έκθεσή σας για το 18 το καταδεικνύει σαφώς. Να πω κάτι από το σοφό Σολομόντα. Λέει Οι πεθαμένες ε, μύγες ε, βρωμίζουν ε, τις αλυφές των θεραπευτών. Οπότε πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να βγάλετε αυτές τις πεθαμένες μύγες. Να μην έχετε αυτές τις δυσχέρειες. Και όπου έχετε τέτοια προβλήματα, να τα αντιμετωπίζετε γιατί η εργασία σας είναι αναγκαία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η συμβολή της ομάδας IND. Ο κύριος Τσαρνιέτσκι από την ομάδα ECR. 1,5 λεπτό. Ε, πρόεδρε, Επίτροπε, Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Ευχαριστούμε το Ελεγκτικό Συνέδριο που πραγματικά έπαιξε έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι ένας σημαντικός ε, θεσμός. Το 2018 οι δαπάνες μας ανήλθαν στα 127 εκατομμύρια περίπου 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό είναι κομβική σημασία αυτές οι δαπάνες να συνάδουν με τους κανόνες να συμμορφώνονται με τους κανόνες. Τα αποτελέσματα, η επίτευξη των στόχων. Αναφέρατε το 2,6% ε, επίπεδο σφαλμάτων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τα ποσοστά που είχαμε τα δύο προηγούμενα έτη. Ε, πέρυσι ήταν 2,4. Ε, το ερώτημά μου είναι ε, αυξάνεται αυτός ο αριθμός, αυτό το νούμερο ή είναι απλώς έτσι μια στατιστική έτσι, διακοσμητική αλλαγή που δεν έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Νομίζω ότι πρέπει να χαιρόμαστε για τις δεσμεύσεις ε, τέλειωσε ο χρόνος μου, οπότε σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο κύριος Φερέιρα για την ΚΟΕ είναι ο ομιλητής, όμως δεν τον βλέπω. Δεν είναι στην αίθουσα. Ε, ο κύριος Χίβερ για 1,5 λεπτό. Η πιο ελαφριά αυτή η έκθεση του ελεγκτικού ε, συνεδρίου έδειξε ότι τα προβλήματα ανέβηκαν. 4,1 ε, δις ευρώ δεν δόθηκαν σωστά τα κονδύλια. Ε, φαίνεται επίσης ότι το τμήμα για το κλίμα που έχει 860 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεση του επειδή δεν έχει καθόλου συναλλαγές, δεν έχει και έλεγχο. Ε, συγκεκριμένη σελίδα που αναφέρεται για στα 9,1 εκατομμύρια ε, που δόθηκαν στις τρίτες ε, χώρες λέτε ότι ο αριθμός των συναλλαγών που ελέγχθηκαν δεν είναι επαρκής για να έχουμε μια εκτίμηση για το επίπεδο σφάλματος. Να σας το πω ξεκάθαρα, δεν θα δώσουμε ούτε δεκαράκι εμείς στη χώρα μου τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τρέχουμε φοβισμένοι και τρομαγμένοι από τις ε, εκλογές, ε, μακριά από τις εκλογές, αλλά δεν μπορούμε να κρυφτούμε για πολύ. Αυτή οι εκλογές θα δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα να σταματήσουν αυτές οι συνθήκες οι οποίες θα μας κάνουν να δώσουμε τόσα χρήματα και να συνεχίσουμε να δίνουμε τα επόμενα χρόνια ή να έχουμε μια ξεκάθαρη απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ξεκάθαρο Brexit και πραγματικά ελπίζω ότι το κόμμα μου θα το πετύχει αυτό στις επόμενες γενικές εκλογές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στεχόφσκι έχει το λόγο. Μα το προφέρατε τέλεια, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτό το τσίρκο το Monty Python είχε τελειώσει εδώ μέσα, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι. Ο κύριος Χίβερ με έπεισε ότι οι Monty Python εξακολουθούν να υπάρχουν και συνεχίσουν τις πολύ πετυχημένες τους παραστάσεις. Κύριε Χίβερ και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας, πραγματικά ενσωματώνεται το πνεύμα των Ponty Python και μάλλον δεν διαβάσατε καν την έκθεση, είχατε δυσκολίες στο να την καταλάβετε. Αναφερθήκατε σε κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες πραγματικά δεν αντιστοιχούν καθόλου στην πραγματικότητα. Αλλά κανείς δεν θα σα κρατάει εδώ πέρα με το ζόρι. Σα το λέω ειλικρινά. Αν θέλετε να φύγετε, μπορείτε να αποχωρήσετε. Αυτό περιμένουμε να μας πει πότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν σας κρατάει εδώ πέρα με το ζόρι τώρα, όσον αφορά την έκθεση αυτή καθεαυτή. Νομίζω ότι αποτελεί ένα θετικό έναυσμα και για άλλους επιτυχημένους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια έκθεση η οποία λέει ξεκάθαρα ότι γίνανε έλεγχοι εξακρίβωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. Ιδίως όσον αφορά κάποια επιμέρους κεφάλαια. Νομίζω ότι θα πρέπει να πετύχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό αποτελεσματικότητος. Πρέπει να δούμε επίσης πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από την έκθεση αυτή, πώς θα στην πράξη τα πορίσματα αυτά της έκθεσης και πώς θα ευαισθητοποιήσουμε για αυτά το ευρύτερο κοινό. Συνολικά λέω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί μια πολύ θετική βάση για τις συζητήσεις που θα πρέπει να κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία πέντε χρόνια πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Και ελπίζω ότι ο κύριος, ο διάδοχος μάλλον του κυρίου, μάλλον ο κύριος Χάντ θα δεχθεί τον κύριο Έτιγκερ, θα εφαρμόσει όλες αυτές τις προτινόμενες εδώ πέρα συστάσεις. Ευχαριστώ κύριε Σδεχόσκη. Δέχεστε από τον συνάδελφο Ρόλαντ μια μπλε κάρτα. Παρακαλώ. Καταρχάς, να συγχαρώ τον συνάδελφό μου. Βλέπω ότι το στηρίζουν πάρα πολύ εδώ μέσα. Καλό είναι να βλέπουμε πόσοι πολλοί τον χειροκροτούν. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Είπατε ότι είμαστε σαν του Monty Python. Πολύ καλή η αναλογία στη ζωή του Brian. Ο κύριος Κρύος δεν ήταν που έφαγε όσο φάει μπορούσε να φάει και νομίζω ότι είναι πολύ καλή η αναλογία με τον προπολογισμό που τρώει όλο και περισσότερα τα πάντα, σουβλάκια, ό,τι να είναι. Δεν είναι σωστή αναλογία αυτή. Καταφέρατε να θέσετε το, την ερώτησή σας σε 31 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Αγαπητέ συνάδελφε, θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά που λέτε, χρησιμοποιώντας μια άλλη παρομοίωση. Την εξής. Συνεχίζεται βεβαίως η Μόντι Πάθρα αλλά και το Yes Minister. Αυτή η τηλεοπτική σειρά. Η ερώτησή σας νομίζω δεν έχει καμία έννοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχει περάσει η ώρα, μόνο μία μπλε κάρτα. Νομίζω ότι όλοι κάνετε την πλάκα σας και η Γκαρθία Μουνιώθ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Έτιγκερ και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρόεδρο Λένε για την παρουσίαση της έκθεσης ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου ως σκιώδης της ομάδας μου για την απαλλαγή προς τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να πω ότι στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου αυτό που δεν είδα ήταν περισσότερα για την οικονομική χρήση των ίδιων. Το 2018 πολύ λίγα λέγονται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Αλλά αυτό είναι όλο. Το ποσοστό σφάλματο βεβαίω ήταν πολύ χαμηλό τα τελευταία χρόνια. Αλλά είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο για τι λειτουργικές δαπάνε των άλλων ε, οργάνων. Θέλουμε να γίνονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο, με περισσότερη αυστηρότητα. Έτσι θα βοηθήσουμε και το Κοινοβούλιο να ελέγξει τι δαπάνε του. Εφόσον την ε, κάνει αυτή την εργασία και κάνει μια αιτήσια έκθεση για κάθε ένα από του εξωτερικού θεσμού, του 41, πιστεύω ότι θα είχε τα μέσα και το προσωπικό και του πόρου να κάνει μια έκθεση και για τα 8 θεσμικά όργανα τη Ένωση, τα κύρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπουαγέ, Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Σα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, την εποπτεία αυτή του κοινοτικού προπολογισμού. Όπω είπε, ο προπολογισμό αυτό αντιστοιχεί στο 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματο, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε κυρίως εισφορές κατά το 80% από τα κράτη-μέλη που κατανέμονται τη συνεχεία στα διάφορα προγράμματα, ένα σύστημα το οποίο είναι πολύπλοκο και το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν οι πολίτες και οδηγεί πολύ συχνά στον εύκολο λαϊκισμό, το είδαμε αυτό και στο μεκύκλειό μας. Η φυστάμενη πολιτική κατάσταση βέβαια μα αναγκάζει αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πλέον ένα προπολογισμό ο οποίο θα βρίσκεται στο ύψο των φιλοδοξιών τη, ένα προπολογισμό ο οποίο θα τροφοδοτείται πλέον από του ιδίου πόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί επιπλέον φορολογία που να βαρύνει τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε βέβαια και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να έχει τα δικά της προγράμματα, τα δικά της έργα, τα οποία να προωθούν πραγματικά το ευρωπαϊκό συμφέρον πανευρωπαϊκά. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά τους ψηφοφόρους μας στις επόμενες εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να εμφυσίσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πολίτες απέναντι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, συνάδελφος Λεμπρετό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Εθνική Συνέλευση θεωρούσε πάντοτε ότι η πολιτική του ασύλου έπρεπε να είναι εθνική πολιτική την δικαιώνει η έκθεση του ελεγκτικού ε, συνεδρίου το 2019 που αναφέρει τα σκανδαλώδεις δαπάνες ε, στο ε, θέμα του ασύλου. Εκεί συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το γραφείο που ασχολείται με το άσυλο έχει υπογράψει συμβόλαια 3,5 εκατομμύριων ευρώ. Το 2018 είχαμε 50 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν για παράνομους σκοπούς. Ε, είναι τόσο κατάφορη αυτή η παρανομία που δεν μπορούμε να μην τη δούμε. Επίσης ε, φαίνεται ότι υπάρχει εκθετική αύξηση των ε, δαπανών σε σημείο που έπρεπε ο Γενικός Διευθυντής να απαρατηθεί. Πολύ καλά κάνει λοιπόν τη δουλειά, της, τη δουλειά του το ελεγκτικό συνέδριο, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει την πολιτική ασύλου πίσω στα κράτη-μέλη. Η συνάδελφος, Η για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Λένε και τον κύριο Επίτροπο. Μας υπέβαλαν μια έκθεση μεγάλης αξίας για να κατανοήσουμε τους λογαριασμούς της Ένωσης. Όπως είπαν και οι δύο, το 2018 τα σφάλματα συνολικά για τις δαπάνες ήταν κάτω από το 2,4%. Είναι προφανές ότι έγιναν προσπάθειες για να μειωθούν τα σφάλματα που πρέπει να συνεχιστούν και συγκεκριμένα για την κοινή γεωρική πολιτική. Ξέρω ότι γίνεται προσπάθειες ε, απλούστευσης ε, του έργου των ε, εθνικών διοικήσεων. Αλλά παρόλα αυτά αυξάνεται για τον τελικό δικαιούχο η πολυπλοκότητα, που είναι φυσικά η γεωργή. Η έλλειψη η απλούστευσης, η γραφειοκρατία που όλο και θεριεύει και η πολυπλοκότητα των εντύπων που πρέπει να συμπληρώσουν Όλα αυτά περιπλέκουν τη δραστηριότητα των εργατών μα. Δεν του μένει χρόνο στο, για το χωράφι. Ελπίζω το ελεγκτικό συνέδριο να συνεχίσει να απαιτεί από την Κομισιόν καλύτερο συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η επόμενη, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, η συνάδελφο Πινιέντολη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για το έργο του. Η αιτήσια αυτή έκθεση είναι ένα κείμενο πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί διευκολύνει τη δική μα την εργασία, μα δίνει πάρα πολλέ πληροφορίε για, να αξιο... αξιολογήσουμε τι δαπάνε από τον κοινοτικό προπολογισμό, να τοπίσουμε και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Στην αιτήσια αυτή έκθεση του 2018 είδαμε κάποιε βελτιώσει σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Πρώτον, εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι το επίπεδο σφάλματο για τι καταβληθεί στι δαπάνε έχει μειωθεί. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα προ σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειε για περισσότερη διαφάνεια χρησιμοποιώντα του δημόσιου πόρου και παράλληλα θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με το λεκτικό συνέδριο. Υπάρχουν κάποια επικριτικά σημεία για το κεφάλαιο 3. Εκεί πέρα επαναφερόμαστε ε, στι πολιτικέ όσον αφορά τον πολίτη, καθώ επίση και στον τομέα 4, η Ευρώπη στο παγκόσμιο προσκήνιο. Δεν καταφέραμε να μειώσουμε το επίπεδο σφάλματος. Υπάρχει ένα μειωμένο επίπεδο διαφάνεια. Για παράδειγμα, η συνοχή κυρίω στι αγροτικέ περιοχέ δεν μα δίνει πάρα πολλέ πληροφορίε και επίση δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε όσον αφορά τα προγράμματα όπω το Εράσμου. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα προβλήματα αυτά το στομότερο δυνατό. Καλύτερη λοιπόν οργάνωση των ελέγχων πρέπει να έχουμε. Να αυξηθούν οι επιθεωρήσει προκειμένου να εξακριβώσουμε τελικά αν τα προγράμματα και οι πολιτικέ υλοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό και αν τελικά τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου πιάνουν τόπο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναλυφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχο αυτό προ το συμφέρον των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξοπιστία του. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό η συνάδελφο Νόβακοφ. Ο συνάδελφο Νόβακοφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, να πω ότι εκπλήσωμαι τόσο πάθος εδώ σε αυτή την παρουσίαση της έκθεσης του ελεγκτικού ε, συνεδρίου. Δεν το περίμενα. Καλό είναι που το βλέπουμε. Υπόθηκαν πολλά για τα νούμερα, τις στατιστικές και τα ποσοστά στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και σωστά. Θα ήθελα όμως να δω τι γίνεται πίσω από τους αριθμούς. Τα άτομα τις εταιρείες, τα project. Είναι καλό που ψάχνετε ποσοστά σφάλματος. Είναι η δουλειά του. Είστε, είναι η δουλειά σας και είστε ο καλύτερος φίλος των φορολογούμενων. Όμως όταν ψάχνουμε τα σφάλματα σε ένα project θα πρέπει να κοιτάμε και τη γενικότερη ποιότητα του project, του έργου. Δηλαδή, έφτασε στο στόχο που επεδίωκε. Έγινε αυτό με το σωστό τρόπο. Δεν πρέπει λοιπόν να κοιτάμε μόνο πώς ε, δαπανήθηκαν οι πόροι, αλλά και πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ένας από τους λόγους που απορροφήσαμε μόνο το 30% των πόρων ε, και για πέμπτη συνεχή χρονιά είναι η γραφειοκρατία. Υπάρχει ο έλεγχος βάση κινδύνου. Αυτοί οι ωφελούμενοι που ε, ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν τα κονδύλια πρέπει να ελέγχονται λιγότερο. Αυτοί που συνεχώς διαπράττουν σφάλματα χρειάζεται να ελέγχονται περισσότερο. Μόνο έτσι θα βρούμε μια ισορροπημένη λύση για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των φορολογούμενων και για να ενθαρρύνουμε τους ωφελούμενους να συνεργαστούν μαζί μας. Ευχαριστώ και τώρα για ένα ε, λεπτό η συνάδελφος Τσινίτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ετήσια έκθεση για το 2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου μα παρουσιάζει μια οικονομική κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι βελτιωμένη σε σχέση με τα παρελθόντα έτη, μολονότι ακόμα υπάρχουν κάποιοι τομεί όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν παρατυπίες και σφάλματα, ιδίω όσον αφορά τι δαπάνε υψηλού κινδύνου, κυρίω για το Ταμείο συνοχή και για την κοινή γεωργική πολιτική. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είπε ότι η πολυπλοκότητα πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια οδηγεί από μόνη τη σε σφάλματα. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια πρόσβαση κυρίω για του μικρού επιχειρηματίε και του γεωργού, οι οποίοι να είναι πιο απλουστευμένοι και να μην κάνουν εσφάλματα κατά αυτόν τον τρόπο. Και όσον αφορά την πρόληψη, μόνο 11 κράτη-μέλη έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά της απάτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει μια καλύτερη ομοιογένεια διοικητική και οργανωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε κοινέ πολιτικέ κατά της απάτης, καθώς επίσης και προληπτικές πολιτικές και πολιτικές για μια καλύτερη παρακολούθηση και εποπτεία του κοινοτικού μας προπολογισμού. Επόμενη για ένα λεπτό η συνάδελφος κυρία Γιούτσικα. Ο συνάδελφος κύριος Γιούτσικα. Ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο για την εξαιρετική δουλειά. Εδώ και χρόνια το συνέδριο ε, πραγματικά έχει εξετάσει προγράμματα και έχει δει τις επιθώσεις, ε, την απόδοση ε, των project σε συνδυασμό με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μας έδωσε επίσης μια εικόνα για τους στόχους ε, που πετυχαίνονται με την ευρωπαϊκή αυτή χρηματοδότηση. Το ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός ως στόχο δεν πρέπει να έχει το να παίρνουμε τα χρήματα από τη μια τσέπη και να τα βάζουμε στην άλλη. Πρέπει το κάθε επενδυθέν ευρώ να φέρνει τα μέγιστα δυνατά ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό ακριβώς ε, το στοιχείο μας έδειξε το ελεκτικό συνέδριο αυτό ε, φαίνεται και στην τελευταία μελέτη του ΟΣΑ όπου αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις περισσότερες πληροφορίες για τον ε, προϋπολογισμό. Είναι στην πρώτη θέση λοιπόν και ειδικά για τα hard data όμως ε, βρισκόμαστε στην τελευταία θέση. Ευχαριστώ. Δεν μπορούμε τώρα να ξεπερνάμε το χρόνο μας πάνω από 50%. Συγγνώμη. επόμενο ε, για ένα λεπτό ο συνάδελφος Μόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν καθώς ε, διέσχιζα το σαλόνι μου, άνοιξα την τηλεόραση και για άλλη μια φορά άκουσα για την ε, πόσο γεννόδορη είναι η Ευρώπη. Όμως ε, ε, πάντοτε πρέπει κανείς να βλέπει την καλή πλευρά. Φεύγουμε από την Ευρώπη και με λένε και Μπράιαν. Στην προηγούμενη ζωή του Μπράιαν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Σκοτσέζικου Κοινοβουλίου για τέσσερα χρόνια και αυτά τα νούμερα εμένα δεν με ξεγελούσαν. 2,6% ε, λάθη σημαίνει 4 δις ευρώ. 4 δις είναι ε, περισσότερα από όσα δίνουν κάποια κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σκεφτούμε τους στόχους, ας πούμε, το να πληρώνουμε τις πτήσεις προσωπικού στη Τζαμάικα με έναν προϋπολογισμό που χρηματοδοτεί τη Ρίβαν.